Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση Ντεκεζέρ για την ανάπτυξη και την οικοδόμηση κράτους στο Νότιο Σουδάν. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ντεκεζέρ για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ κυρία Ντεκεζέρ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την έκθεση τους σκιώδει εισηγητές αλλά και τους συναδέλφους από τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπές που έδωσαν πολύ εύστοχε απόψει, ιδίως από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Το Νότιο Σουδάν είναι το τελευταίο κράτος στην Αφρική που απέκτησε την ανεξαρτησία του εδώ και τρία χρόνια, τον Ιανουάριο του 2011. Έγινε αυτό με ένα δημοψήφισμα και τον Ιούλιο του 2011 ανακηρύχθηκε επισήμως στις 9 Ιουλίου η ανεξαρτησία του. Μετά από πέντε ημέρες, το... η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δέχτηκε τον Νότιο Σουδάν ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, η ταχύτητα αυτή <clears throat> δεν ήταν τυχαία γιατί αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό από όλη τη διεθνή κοινότητα μετά την συνθήκη ειρήνης του 2005 που έθεσε τέρμα σε ένα ατέλειωτο εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν που είχε επιπτώσει σε όλη την γειτονική περιοχή. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο, έχουμε ένα νέο κράτος, το οποίο βέβαια είναι ένα έφραστο κράτος, έχει πετρελαϊκούς πόρους, αλλά μόνο πετρελαϊκούς πόρους. 90% της οικονομίας του στήριζεται στο πετρέλαιο αλλά έχει ένα μεγάλο γείτονα, το Σουδάν, όπου δεν έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις από τη στιγμή που υπήρξε η απόσχηση του Νοτιού Σουδάν. Εδώ και τρία χρόνια μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις, διακοπή της κυκλοφορίας του πετρελαίου που θίγουν και τη μία και την άλλη χώρα και η διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τρόικα όχι η δική μας Τρόικα, είναι η Τρόικα που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, Μεγάλη Βρετανία και η Νορβηγία. Έχει δημιουργήσει φόρουμ όπως αυτά στην Ουάσιντον για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει να υπάρξουν <clears throat> κάποιες ε, βελτιώσει την κατάσταση του Νοτιού Σουδάν και να αποτρέψουν την χρεοκοπία της χώρας αυτής. Αυτή τη στιγμή 50% του πληθυσμού του Νότιου Σουδάν βρίσκεται κάτω από το κατόφλι της Ένδειας. <clears throat> Είναι απόλυτη η εξάρτηση της χώρας αυτής από το πετρέλαιο, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η συμφωνία της Κοτονού δεν έχει ακόμα ε, υπογραφεί από τον Νότιο Σουδάν. Είναι δύσκολο λοιπόν να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει διαδεδομένη διαφθορά η οποία είναι ενδημικού χαρακτήρα, είναι πολύ ψηλό το ποσοστό παιδικής και μητρικής συνσημότητος, 48% των ε, νέων γυναικών ε, παντρεύονται μεταξύ σε ηλικία που δεν ακόμα ενήλικες ε, εναντίον της θέλησης περισσότερες φορές. Υπάρχουν πολιτοφυλακές που δεν είναι μέσα στις στένοπλες δυνάμεις, υπάρχουν ληστείες, φόνοι, βιασμοί, καταδιώξεις των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα <clears throat> πραγματικό πρόβλημα ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπάρχει μια νομοθεσία η οποία είναι στα αγγλικά, ο πληθυσμό δεν καταλαβαίνει μία. <clears throat> Εάν αυτή η χώρα όμως αποτύχει, όλη η περιοχή του κέρατος της Αφρικής θα αποσταθεροποιηθεί για μια φορά ακόμα. Εδώ υπάρχει μια παράγραφο στο ψηφισμά μας που συνοψίζει τις ε, προτάσεις μας για να επιτευχθεί μια καλή διακυβέρνηση και να υπάρξει ένας αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νέο. Το Νότιο Σουδάν είναι η παράγραφος 9, καθώς και η παράγραφος 11. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές, <clears throat> γιατί το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 830 εκατομμύρια για τον Νότιο Σουδάν. Πολλά λεφτά, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Και Πολύ σπάνια αναφέρεται το θέμα αυτό. Είναι μια χώρα η οποία πρέπει να αποκτήσει δημοκρατικές δομές, θα πρέπει να συνεχίσουμε να την βοηθούμε, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερες υποδομές, καλύτερη παιδεία, καλύτερη διακυβέρνηση και να βρεθούμε μαζί με τον Νότιο Σουδάν, αλλά να τους βοηθήσουμε να φτάσουμε μια διακυβέρνηση η οποία να μην διατρέχεται από την διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ε, ο κύριος Στίερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτήν την πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε σχετικά με την έκθεσή του. Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αναπτυχθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ ε, του Νοτίου και του Βορείου ε, Σουδάν Γνωρίζουμε ότι η οικονομία του Νοτίου ε, Σουδάν ε, βασίζεται στο πετρέλαιο, αλλά βεβαίως ε, αυτό το πετρέλαιο θα πρέπει να προωθηθεί προς τον Βορρά. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη τι πολύ κακέ σχέσει ανάμεσα στα δύο, στις δύο ε, αυτέ χώρε, Βόρειο και Νότιο Σουδάν, θα πρέπει η, Ευρωπαϊκή Δημοπλα... <clears throat> διπλωματία να παίξει σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές ε, διότι η επιδείνωση των σχέσεων των δύο αυτών ε, χωρών θα ε, δημιουργήσει προβλήματα σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία ήδη έχει αναφέρει η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Uh, it's not that long ago when we discussed uh, South Sudan. Δεν είναι πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα στα κατεπήγοντα της πέμπτης το απόγευμα και ειδού το ξανασυζητούμε σημάδι της προσήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση του Σουδάν σε αυτήν την ε, ευάλωτη περιοχή σε αυτό το εύθραυστο νέο κράτος το λέω διότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και πρέπει να βοηθήσουμε και εμπροκειμένο. Υπάρχουν δυνατότητες στην περιοχή που δεν έχουμε αξιοποιήσει. Υπάρχουν δυνατότητες ε, βάσει των φυσικών πόρων, για παράδειγμα. Χρειάζεται όμως η απαραίτητη υποδομή ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί. Η χώρα αυτή έτσι θα γίνει πιο ανεξάρτητη και πιο βιώσιμη. Και βεβαίως το θέμα της παιδείας, ζωτική σημασία για όλους. Πρέπει να διορθώσουμε την στάση επένδυση στην παιδεία και ειδικά την εκπαίδευση των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι γραμμένοι αγορητέ και επομένω η κυρία Ντεκεζέρ να απαντήσει. Παρακαλώ, κυρία Ντεκεζέρ. Όχι, δεν θέλει. Επομένω θα δώσω αμέσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ. Παρακαλώ, κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω και να επενέσω την κυρία Ντεκεζέρ, όχι γιατί εκπώνησε μια εξαιρετική έκθεση αλλά και γιατί η έκθεση αυτή προέκυψε μέσα από μια μεγάλη διαδικασία προετοιμασίας ε, και διαβουλεύσεων. Πρόκειται εδώ για μια χώρα η οποία ε, ε, ταυτοχρόνως ε, μας δίνει το μέγεθος των προβλημάτων αλλά και το μέγεθος των προκλήσεων και των δυνατοτήτων ε, πολλά σημαντικά σημεία αναφέρονται στην έκθεση αυτή που μπορεί να αποτελέσει οδικό χάρτη για την, ε, όχι μόνο για, για τον Νότιο Σουδάν αλλά και για την αντιμετώπιση ολόκληρης της περιοχής. Δεν μπορεί κανείς ε, να καταλάβει πραγματικά την οικονομική κατάσταση αν δεν λάβει υπόψη κάποια ιστορικά στοιχεία ε, αν δει κανείς όμως τι κατάφερε η χώρα αυτή μέσα σε 8 χρόνια, ε, πώς μπόρεσε να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών της ε, στην εκπαίδευση, δημιούργησε καλύτερες συνθήκες ευζοίας, βελτίωσε το θεσμικό πλαίσιο, πραγματικά θα μείνει κατάπληκτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως τα μάλα υποστήριξε την χώρα αυτή και τις προσπάθειες που έχει καταλάβει, καταβάλει, συγγνώμη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει περαιτέρω να στηρίξουμε και την κοινωνία των ε, πολιτών. Εμείς ε, είμαστε πλέον σε συνεργασία με τους κυριότερους ε, παγκόσμιους παίκτες και επομένως νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλαίσια αμοιβαίας λογοδοσίας. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να εφαρμοστεί και η Συμφωνία της Κοτονού έτσι ώστε να μπορέσουν να οικοδομηθεί μια μακρόχρονη ε, εταιρική ε, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τον ρόλο των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών στη διαδικασία επούλωσης των πληγών ε, η εξαίρεση, ο αποκλισμός των γυναικών και των κοριτσιών από την ενεργή ζωή ε, είναι μια συστημική δυσκολία η οποία δημιουργεί ένα μεγάλο φραγμό στην ολοκλήρωση της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση Swinburne σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση για μη πιστοτικά ιδρύματα.